ψηφοφορία για αυτή τη συζήτηση θα γίνει στις 12 η ώρα. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ευαισθητής διατάξεως. Πρόκειται για την υπόθεση του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου Σέσελη. Και θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ιγνάτζιο Κοράου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο υπερεθνικιστής ε, ηγέτης ε, του κινήματος ε, για την απελευθέρωση της Βόρειας Σερβίας επέστρεψε στο Βελιγράδι πριν από λίγο καιρό και εκεί ε, στο Βελιγράδι διοργανώθηκε ε, μια εκδήλωση πρόκειται για έναν άνθρωπο που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου όμως ε, οι πολιτικοί δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο πόλεμο και στα εγκλήματα. Το θέμα στο οποίο ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ στη Σερβία ήταν η απόφαση του δικαστηρίου της ε, Άγης αν έχει το δίκαιο για τον Σεσέλ και αν μπορεί να εξυπηρετήσει τους Σέρβους. Ο Σεσέλ κινήθηκε πολύ ωραία χωρίς τη βοήθεια κανενός, μάλιστα έκανε ομιλίες πολιτικού ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί να κοιτώντας ε, για έναν μύθο, έναν μύθο που δίθεν διέπραξε εγκλήματα ε, εναντίον της ανθρωπότητας ε, υπάρχει κίνδυνος για πολύ αθέμητες καταστάσεις. έτσι. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω πλήρως αυτό το ψήφισμα και την επικριτική προσέγγιση όχι μόνο προς τον Σέσελη αλλά και όσους το καταστούν δυνατό ε, για καθημερινά να συνεχίζει τη... το λόγο μίσους για την προπαγάνδα για την Μεγάλη Σερβία. Ολόκληρο αυτό το, το τσίρκο δεν θα υπήρχε αν οι σερβικές αρχές αμέσως είχαν απομακρυνθεί και είχαν κατα καταδικάσει αυτές τις έξι δηλώσει, τι οποίες προέβη ο Σέσελη. Ξέρω πως ήμασταν συνάδελφοι στο παρελθόν και στενοί συνεργάτε, όμως τώρα είναι ηγέτες της ε, Δημοκρατία τη Σερβίας και είναι προ το δικό του συμφέρον να τον συλλάβουν και να τον καταδικάσουν και να προχωρήσουν προς την Ευρώπη. Πραγματικά με εντυπωσιάζει η έλλειψη αποτελεσματικότητας του δικαστηρίου που δεν έπαιξε τον ιστορικό του ρόλο, αντίθετα οδήγησε σε μεγαλύτερη διχόνοια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σκυρλέκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προχτές ο Πάπας μίλησε στο Κοινοβούλιο και μας είπε πως θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα μίση του πολέμου ο Σέσελη όμως προσβάλλει τη συλλογική μνήμη των ε, Κροατών πολιτών παρά το ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γνώριζε τους κινδύνους, έδρασε ανεύθυνα και έτσι μπορεί να αποσταθεροποιηθεί η περιοχή και βεβαίως και το όργανο αυτό αναμένο από τα θεσμικά όργανα της Σερβίας να δράσουν υπεύθυνα όπως αρμόζει σε μια υποψήφια χώρα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, οι καλές γειτονικές σχέσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στηρίζω τα πολιτικά κόμματα και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών στην Σερβία στην προσπάθειά τους να επιτύχουν μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Είμαι σίγουρος πως ε, στον δρόμο της για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία θα κάνει αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτό το ψήφισμα. Βάιντεν Χόλτσερ για ένα λεπτό. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Το παλθόν ρίχνει τη βαριά σκιά του στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τα εγκλήματα δεν ε, μπορούν απλά, δεν μπορούμε απλά να τα σπρώξουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονικές δικαστικές διαδικασίες, να εξακριβωθεί η αλήθεια, κάτι το οποίο συχνά διαρκεί πάρα πολύ, όπως στην περίπτωση Βόησλαβ Σέσελη. Το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο προσωρινά για ανθρωπιστικούς λόγους όπως συνηθίζεται στα κράτη δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για μελλοντικέ αποφάσεις. Και δεν είναι δυνατόν η περιοχή να ζει συνεχώς στο παρελθόν. Πρέπει να γίνονται σεβαστά ε, τα να γίνονται σεβαστοί οι θεσμοί της δικαιοσύνης. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν έτσι οι λαοί της περιοχής όσο δεν αντιμετωπίζουν το παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ράντος για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την απελευθέρωση του Σέσιλι δεν ήταν σωστή και επίσης βεβαίως πρέπει να καταδικάσουμε την επίθεσή του στη Βοσνία και την Κροατία. Ο Σέσελη είναι άρρωστο, άλλοι λένε πω είναι και τρελό. Είναι, εν πάση περιπτώσει, εγκληματία πολέμου. Δεν θα του αλλάξουμε τι απόψει. Και, και το Διεθνέ Δικαστήριο για τη Ιουγκοσλαβία ούτω ή άλλω πλησιάζει στο τέλο τη θητεία του. Η Σερβία τώρα είναι το θέμα μας εδώ πέρα γιατί η μοίρα άλλων χωρών της Βαλκανικής εξαρτάται από την Σερβία και μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα θετικά ή αρνητικά. Γι' αυτό πρέπει να καταδικάσουμε αυτά τα οποία είπε ο Σέσελη, την επίθεσή τους γειτονικές χώρες και ακριβώς πρέπει να ενισχύσουμε τους νόμους που απαγορεύουν ε, το κήρυγμα μίσους και υποστηρίζουν την βία. Μαρή Κριστίν για ένα, Βερζιά για ένα λεπτό. Δεν δε, δε, χρειάζεται να αναφέρουμε όλα τα ελληνικά για τα οποία κατηγορείται ο κύριο ε, Σεσέλη. Ε, είμαστε τι είχε πει ο, ο, ο Μιλόσεβιτ και είναι πρώτο για τους έθνες, τους δεξιούς και είδατε τι έκαναν τότε με τους Ναζί στο δεύτερο πόλεμο και υπήρξε καταδίκαση, καταδίκη από το Χάγη, το δικαστήριο της Χάγης 15 μήνες αλλά ακόμα δεν έχει δικαστεί για τα κυριότερα εγκλήματα και για λόγους υγείας απελευθερώθηκε, πήγε στη χώρα του πίσω και ξανά να τη γλώσσα του μίσους. Οπότε τα θύματα του δικαιούνται να αποδοθεί δικαιοσύνη, θα πρέπει να καταδικαστεί και έτσι ε, θα φέρουμε την ε, συμφιλίωση. Το χρειάζεται αυτό η Σερβία. Ε, όμως ε, ήδη χρησιμοποιεί το κείμενο αυτό του ΕΛΚΑ η πλευρά του τόσο ώστε να, να είναι στη δημοσιότητα οπότε θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη επιλογή των κατεπηγόντων να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού σε όλο τον κόσμο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Με αυτό το ψήφισμα προβαίνουμε στην κατηγορηματική καταδίκη της γλώσσας του μίσους που χρησιμοποιεί ο Σέσελ από το που γύρισε στο Βελιγράδι. Θα πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή της στο δικαστήριο της Χάγης. Θα πρέπει να τον καταδικάσει Καταδικάζουμε τη γλώσσα του μίσους γιατί έχουμε τόσα θύματα ε, τόσους Κροάτες που σκοτώθηκαν στο Βούκοβαρ. Θα πρέπει να μην ανοίγονται νέες πληγές και επίσης θα πρέπει να σταματήσουν οι νέες εδαφικές βλέψεις της Σερβίας που θα τη φέρουν σε σύγκρουση με, τους, με τις όμορες χώρες. Θα έπρεπε αλλιώς να αντιδράσουν σε ελληνικές αρχές, όχι αυτό το οποίο έκαναν. Να κάνουν κάτι άλλο. Και επίσης ο Σέσιλ έχει παραβεί και το σερβικό δίκαιο. Θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προς την Σερβία ότι πρέπει να καταδικάσει τον Σέσελη. Ο πρόεδρος Βούτσιτς και ο πρόεδρος ε, Νίκολιτς ίσως φοβούνται η σιωπή τους δημιουργεί υποψίες. Θα πρέπει η Σερβία κάτι κάτι να αντιδράσει και να δικάσει τους εγκληματίες πολέμου. Ο επόμενος. Πρόεδρε, καταλαβαίνω ακριβώς το τι γίνεται με αυτού του είδους ε, τη γλώσσα του μίσους, πόσο, πόσο θέτει σε αμφιβολία την ε, ευάλωτη ειρήνη των ε, Βαλκανίων. Επομένως, ακριβώς γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί θα πρέπει να έχουμε μία αντίδραση η οποία όμως να μην φέρει περισσότερη ένταση. Δεν θα πρέπει αυτός ο εγκληματίας πολέμου να ελκύει την προσοχή. Δεν το αξίζει. Αυτού του είδους οι ριζοσπαστικές δηλώσεις του Σέσελη ε, ήλκησαν τα, τα, μέσα ενημέρωσης, ε, πολύ πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει όλα αυτά να φέρουν περισσότερη πολιτική ένταση στην περιοχή. Ούτε το ψήφισμα είναι ο κατάλληλος τρόπος να υπαγορεύσει κανείς το τι θα κάνει το ε, Διεθνές Δικαστηρίο. εντολή του είναι ξεκάθαρη. Γι' αυτό και εγώ διστάζω να επιψηφίσω το κείμενο. Ένα λεπτό, πίτσουλα. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια κατάσταση εξαιρετικού χαρακτήρα. Έχουμε ε, μια κατάσταση η οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Να μην θεωρείται αυτονόητη η σταθερότητα και η ειρήνη στα Βαλκάνια. Χρειάζεται κατεπηγόντως να καταδικαστεί ο Σέσελιο. Δεν έχει μετανοήσει για όσα έκανε ο Σέσελιο όλες αυτές τις πληγές που δημιούργησε στα Βαλκάνια. Η προσωρινή του αποφυλάκηση οδήγησε στο να ξανανοίξουν οι πληγές που είχαν ανοίξει την δεκαετία του 90. Θα πρέπει οι σερβικές αρχές να διαπιστώσουν κατά πόσον ο Σέσελη παρανόμησε και παρέβη το σερβικό δίκαιο. Δεν μπορεί να διαδίδει όλες αυτές τις ιδέες που κόστησαν τόσο πολύ στην Σερβία και στις ε, γειτονικές χώρες. Председател, уважаеми ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ πλήρως με τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτό το ψήφισμα. Το όνομα του Σέσελη σημαίνει εγκληματίας πολέμου. Είναι σύμβολο του εμφυλίου της Ιουγκοσλαβίας ε, που μενόταν για πάνω από 10 χρόνια κατέστρεψε τις ζωές ε, ανθρώπων, ε, κατέστρεψε σπίτια, κατέστρεψε τις ε, σχέσεις στα Βαλκάνια και κατέληξε στον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Συνεχίζει αυτή η πολιτική, αυτά τα οποία έκανε στο Σέρεμπροτς και αλλού. Δεν μπορούμε απλά να καθόμαστε. Έτσι, οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να είναι στη φυλακή. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Βάγγελ. Ε, μικρόφωνο παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Ο στα, στην πρώην Ιουγκοσλαβία έχει καταστεί συνώνυμος του εγκληματία πολέμου και με την ε, προσωπικότητά του σημάδεψε τη μάχη του Βούκοβαρ. Το όνομά του θα αναφέρεται μαζί με τους Ναζί και τους φασίστες. Δεν του αξίζει δημόσιο βήμα μιλάει για τις ε, παλιές ιδέες. Τώρα δεν θέλω να ασκήσω κριτική στο δικαστήριο της Χάγης, αλλά δεν ήταν και ευφυής αυτή η απόφαση. Όσον αφορά τώρα την σερβική κυβέρνηση, αποστασιοποιήθηκε και απευθύνω έκκληση στη σερβική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Σόλτες, εγώ συνυπέγραψα αυτό το ψήφισμα. Γιατί, όχι γιατί θέλω εγώ να κρίνω την ευθύνη του, αυτό είναι ευθύνη του δικαστηρίου της Χάγης δεν συνυπέγραψα γιατί δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε μαθήματα στη Σερβία. Η Σερβία έχει αλλάξει πλήρως από την εποχή του Σέσελι. Πριν ακόμα βγει η απόφαση αυτό που γνωρίζουμε είναι πως δεν επιτρέπεται να κάνει αυτά τα κηρύγματα μίσους ο Σέσελη που θα οδηγήσουν σε νέες εντάσεις. Στο κοινοβούλιο αυτό θα έρθουν μία μέρα και οι Σέρβοι συναδελφοί μας και πρέπει οπωσδήποτε να τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο για ένα λεπτό σε λίγη ώρα θα κληθούμε να αποφασίσουμε για, την τύχη του δόκτωρα σέσελη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παραμείνει για 12 χρόνια στη φυλακή ως πολιτικός κρατούμενος όχι για όσα διέπραξε αλλά για όσα είπε δηλαδή για τις ιδέες του. έχετε διανοηθεί ποτέ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να καταδικαστεί ο αρχηγός του κόμματος με το οποίο έχετε κλεγεί χωρίς να έχει διαπράξει αδίκημα. θα μου απαντήσετε όχι γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία. οι έλληνες εθνικιστές όμως δυστυχώς θα σας απαντήσουμε ναι διότι εδώ και δεκατέσσερι μήνε ο αρχηγό έξι βουλευτέ και στελέχη του κόμματό μα βρίσκονται άδικα και παράνομα στη φυλακή όχι διότι διέπραξαν κάτι κακό όχι διότι είπαν κάτι κακό αλλά απλώ επειδή οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με πολιτικά επιχειρήματα τα δικά του επιχειρήματα δικαστική αυθαιρεσία κατόπιν κυβερνητικής εντολής θα μου πείτε και θα συμφωνήσω μαζί σας. δυστυχώς τα δημοκρατικά κράτη όταν το επιβάλλουν πολιτικές σκοπιμότητες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο ίσως και χειρότερο των, ε, κρατών των ολοκληρωτικών τα οποία εμείς καλώς καταδικάζουμε. Ευχαριστώ κύριο Μακάλιστερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το βασικό μήνυμα εδώ πέρα του ψηφίσματός μας είναι να καταδικάσουμε την ερητορία μίσους ε, του κυρίου Σέσελη. Η ενθάρρυνση αυτή εδαφικών διεκδικήσεων δεν έχει θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ενθαρρύνουμε όλες τις σερβικές αρχές, ε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τα πολιτικά κόμματα, νοικιό και όλους τους ανθρώπους να παλέψουν αυτό το κήρυγμα μίσους. Εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω την Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία. Έχει δηλώσει πως η ένταξη είναι στρατηγικός της στόχος και όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει κάνει η Σερβία σαφώς ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να στηρίξουμε τη Σερβία στην προσπάθεια αυτή. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Να πω στους ε, συναδέλφους πως δεν έχουμε χρόνο, οπότε δεν θα δεχτούμε μπλε κάρτες ε, και ζητώ την κατανόησή σας. Ουλιαστόφσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Απευθύνω έκκληση στο δικαστήριο της Χάγης επιτέλους να δικάσει αυτές τις υποθέσεις. Μιλάμε εδώ πέρα πως στο ψήφισμα για εγκλήματα. Μα, για να υπάρχει δικαιοσύνη πρέπει να τιμωρηθούν όλα τα εγκλήματα. Και αυτά που έγιναν επί κομμουνισμού, τα οποία δεν δικάστηκαν. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι πως πρέπει να καταδικάσουμε τον κύριο Σέσελη και τα εγκλήματά του δεν θα πρέπει να κλείσουμε την πόρτα στο μεγάλο σερβικό έθνος που έχει δικαίωμα να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα όπως όλες οι χώρες των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Ευχαριστούμε. Ιβάν Γιακοψίτς για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, το δικαστήριο της Χάγης έχει συσταθεί για να καταδικάσει τους εγκληματίες πολέμου της πρώην Ιουκοσλαβίας. Αλλά δεν έχει καταπολεμήσει τη διάδοση του μίσους. Το ξέρω ότι δεν είναι σωστό να ε, συζητούμε για δικαστικές αποφάσεις, αλλά η απόφαση αυτή δεν θα συμβάλλει ούτε στην ειρήνη ούτε στην ασφάλεια στα Βαλκάνια. Εδώ στο Κοινοβούλιο η καταδίκη του Σέσελη είναι απερίφραστη και σαφέστατη. Θα ήθελα όμως να τονίσω ε, ότι δεν θα πρέπει να υποδαβλίζεται το μίσος. Η Σερβία έχει σε μεγάλο βαθμό γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά ε, και τα αγνοεί. Ε, ο λαός Σερβίας θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δείξει καλή βούληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κριστιαν Πρέντα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. <clears throat> Να καταδικάσω έντονα τι ε, ενέργειε του Σέσελη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για αποτρόπια εγκλήματα πολέμου στην επικράτεια της Βοσνίας Ερχοβίνης και της Κροατίας τον πόλεμο της πρώην Ιουκοσλαβίας. Έχουμε ακούσει τι ε, λόγια μίσους έχει εκφράσει ως τώρα και ξέρουμε ότι έγινε δεκτός ως ήρωα στη Σερβία αφού απελευθερώθηκε για ανθρωπιστικούς λίγους. Βλέποντα όμω τι αντιδράσει από την Βοσνία Ερζεγοβίνη, είδαμε και τον αποτροπιασμό των θυμάτων. Η έλευση του Σασελή άνοιξε παλιέ πληγέ. Πέρα όμως από αυτά, μπορεί να διακυβευτεί και η προσπάθεια που γίνεται για συμφιλίωση στα Δυτικά Βαλκάνια με την παρουσία του εκεί. Η εμπιστοσύνη του κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν ε, αυξάνεται με τέτοιε ενέργειε. Θα καλέσω λοιπόν την τάξη των πολιτικών εθνών στη Σερβία να καταδικάσουν αυτά τα λόγια μίσου. Στη διαδικασία Κατσιά έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί συνάδελφοι και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το έχουμε συζητήσει το θέμα, δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση και ξέρετε ότι στις 12 ακριβώς αρχίζουν οι ψηφοφορίες, οπωσδήποτε. Γιατί ο κόσμος πρέπει να φύγει από το Στρασβούργο κάποια στιγμή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα δώσω το λόγο σε ένα μόνο που δεν έχει μιλήσει ακόμα στο ΚΑΤΣΙΑΙ και σε κανέναν άλλον. Ήδη έχετε μιλήσει ορισμένοι που ξαναζητάτε το λόγο στη συζήτηση. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε έναν και μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Χάν. Παρακαλώ. Uh, Από ό,τι φαίνεται ε, αποσιάζει ο κύριος Χάν μόλις εξήλθε τις αθώσεις. Ο Επίτροπος κύριος Τηλιανίδης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκ μέρους της κυρίας Μογκερίνη θα σας παρουσιάσω το θέμα αυτό. Ξέρω ότι ε, αρκετοί βουλευτές συζητάνε μία επίγουσα συζήτηση σχετικά με το δικαστήριο που δικάζει τον Σέσελη και γνωρίζω και το ψήφισμα που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Όπως γνωρίζετε, το δικαστήριο έλαβε απόφαση για λόγους υγείας. Δεν έχουμε άλλες απόψεις σχετικά με την απόφαση αυτή. Το δικαστήριο είναι ανεξάρτητο διεθνές δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό ευθυνών διαφόρων ατόμων για εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου. Όσον αφορά τον Σέσελ, ανήκει σε ένα καθεστώς ε, ξεπερασμένο και γνωρίζουμε ότι η υπόθεση εναντίον του συνεχίζεται και ότι θα πρέπει να επιστρέψει στο δικαστήριο όταν του ζητηθεί αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά την Σερβία, επικροτούμε τη δέσμευση της χώρας να εργαστεί με, για την προσέγγιση ε, προς την Ευρώπη και η συνεργασία με το δικαστήριο αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος εξ ονόματος ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων και ε, κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στη συνέχεια. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Ιράκ απαγωγές και κακοποίηση γυναικών. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αλλά σας παρακαλώ να σέβεστε απολύτως το χρόνο σας.